So, meine sehr Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είναι κάπως ισχνή η συμμετοχή στην αίθουσα. Αιτιολογείται μάλλον από το ακαδημαϊκό τέταρτο που έχει γίνει πια και εκτιμένο δικαίωμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Συνήθως στην αρχή της συνεδρίασης είναι κάπως περιορισμένη η συμμετοχή, σήμερα περισσότερο από ό,τι άλλη φορά. Πάντως επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον νέο προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών σε θέματα δικαιοσύνης, Υπουργό ε, Δικαιοσύνης της Κύπρου, κύριο Λουκά Λουκά. Και επιτρέψτε μου πριν σας δώσω το λόγο για να ξεκινήσουμε να δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικές με την ημερήσια διάταξη, μια σειρά από τροποποιήσεις που πρέπει να γυρούν οι διορθώσεις καλύτερα, που θα πρέπει να ανακοινώσω στους συναδέλφους. Το θέμα των διαφορών στο σημείο 10 θα το ε, συζητήσουμε το άλλο. Το 6 δεν θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα, το διαγράφουμε. Τα 8 και 9 θα πάνε αύριο το απόγευμα, γιατί δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα ο εισηγητής. Και το 34 του κυρίου Μπερλίνγκουερ θα το συζητήσουμε σήμερα, τα το απόγευμα μετά τις 4.30. Μετά το σημείο 7 της σημερινής διάταξης. Τα έχω σημειώσει και εγώ στην τελευταία μου διάταξη, ίσω είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσει κανεί τι αλλαγέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ξεκινάμε λοιπόν μετά αύριο το απόγευμα στις 3 με την ακρόαση τη κυρία Κονιλάνγκεν για τα θέματα τη ε, ε, ασυλίας. Μετά στα διάφορα θα έχουμε μία, θα γίνει μετά με ψηφοφορία βέβαια, μετά στα διάφορα θα έχουμε μια θα γινει μετα μετα στα διαφορα θα εχουμε μια συζητηση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που από την ε, προηγούμενη εβδομάδα ξέρουμε ότι παραμένει εκρεμές και έχουμε και μία σειρά θεμάτων το 26, το 27 κ. Γκαργάνη που δεν θα μπορέσουμε για λόγους τεχνικούς να συζητήσουμε. Μετά έχουμε την έκθεση του κυρίου Μπαλντάσαρ για την ε, ε, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που για λόγους πάλι τεχνικούς δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν για την ημερήσια διάταξη. Και έτσι πάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω άλλη ανακοίνωση παρά μόνο σα υπενθυμίσω πάρτε μέσα στι κάρτε σα για την ψηφοφορία στην αυριανή συνεδρίαση. Τα πρακτικά τη 30-31η Μαου του 2012, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, επικυρώνονται. Και έτσι τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στον Κύπριο Υπουργό κ. Λουκά, Υπουργό Δικαιοσύνη. Καλώ ήρθατε, σα καλωσόριζω θερμά και παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, συνεχίζοντας το έργο που έχει επιτυχημένα επιτελέσει η Ιδανική Προεδρία. Η Κύπρος αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Το γεγονός αυτό είναι υψίστης σημασίας για εμάς και καθίσταται πραγματική πρόκληση λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και την πολιτική αστάθεια στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η Κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει τις προσπάθειές της στη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης που θα είναι πιο αποτελεσματική τόσο για τους πολίτες της όσο και για τους γείτονες της. Προς επίτευξη του στόχου αυτού σε ό,τι αφορά τον τομέα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ολοκλήρωση και έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης και παράλληλα η διασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών μέσων τα οποία θα συνδράμουν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων προ αυτήν την κατεύθυνση. Προ επίτευξη των στόχων αυτών η Κυπριακή Προεδρία δηλώνει έτοιμη για στενή συνεργασία και διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο. Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και τη σημασία της στενής συνεργασίας των δύο θεσμικών οργάνων, η οποία μπορεί να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία κάθε Προεδρίας η συνεργασία του Συμβουλίου με την Επιτροπή Γιούρι ήταν πάντοτε εξαίρετη και επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη συνεργασία αυτή στα ίδια υψηλά επίπεδα. Προτεραιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις θα συνεχίσουμε το εξαίρετο έργο της Δανικής Προεδρίας και στοχεύουμε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 επί Προεδρίας. Το νομοθέτημα αυτό αποτελεί το θεμέλιο της δικαστικής συνεργασίας στον τομέα του αστικού δικαίου, καθότι θέτει τους κανόνες για την δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Κύριος σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι η άρση των υφιστάμενων εμποδίων για την διασυνοριακή εφαρμογή αποφάσεων. Κρίνοντας από τις επικοδομητικές ε, ανεπίσημες επαφές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι υπάρχει υψηλός βαθμός συναντήληψης και ότι είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας κατά το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης. Θα εργαστούμε σε συνεργασία μαζί σας για να το επιτύχουμε αυτό. Η Κυπριακή Προεδρία θα εξετάσει ως προτεραιότητα την πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού για την διευκόλυνση της διασυνοριακής ίσπραξης οφειλών. Στόχος είναι να εργαστούμε σκληρά για την επίτευξη τόσο του όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πρόοδου. Ο προτινόμενος κανονισμός είναι πολύ σημαντικός. Θα αποτελέσει το πρώτο νομοθέτημα που θα εισάξει μέτρο εκτέλεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα αυτή προσέγγιση η πρόταση αναμένεται να συμπληρώσει παραδοσιακά νομικά εργαλεία επί της αμοιβαίας αναγνώρισης όπως είναι ο κανονισμός Βρυξέλλες 1. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να προβλεφθεί το κατά πόσο μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση της πρότασης. Αν ληφθούν υπόψη τα δύσκολα θέματα που εγείρονται, το ότι είναι η πρώτη φορά που συζητείται πρόταση για διασυνοριακά μέτρα εκτέλεσης, αλλά και το γεγονός ότι οι συζητήσεις επί της πρότασης βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να προχωρήσει με τις συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας με στόχο την κατάληξη σε μια ολοκληρωμένη πρόταση που να εξυπηρετεί τους σκοπούς της διευκόλυνσης εκτέλεσης απόφασης με την παγωποίηση τραπεζικού λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο αλλά και η οποία θα διασφαλίζει επαρκώς τόσο τα δικαιώματα των διαδίκων όσο και τα δικαιώματα τυχόν τρίτων ατόμων τα οποία δυνατόν να επηρεάζονται από τη διαδικασία αυτή. Προεδρία σκοπεύει περαιτέρω να συμβάλλει στην ενίσχυση της άσκησης των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών, συνεχίζοντας τις εργασίες της δύο προτάσεις κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων. Οι δύο αυτές προτάσεις αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία και πρόθεση μας είναι όπως εργαστούμε εντατικά καθότι θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των δύο αυτών προτάσεων θα διευκολύνει την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Όπω αντιλαμβάνομαι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται το στόχο μα αυτό. Αξίζει να αναφέρω επίση ότι για τα θέματα αυτά θα, πραγματοποιήσουμε συνέδριο στι 9 Οκτωβρίου στη Λευκοσία του 2012 κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Η Προεδρία θα εργαστεί επίση για την υιοθέτηση του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασία σε αστικέ υποθέσει. Η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες εφόσον θα ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων παρέχοντας ένα γρήγορο και εύκολο μηχανισμό διασυνοριακής αναγνώρισης των μέτρων για την προστασία των ατόμων αυτών. Υπάρχουν ακόμη κάποια τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Παραδείγματο χάρη η ακριβή σχέση μεταξύ του προτινόμενου κανονισμού και άλλου σχετικού και χτυμένου, ιδιαίτερα του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και η πρακτική λειτουργία του μηχανισμού αναγνώρισης. Όμως, η Κυπριακή Προεδρία, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η πρόταση αυτή για τα θύματα, στοχεύει στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Όσον αφορά την προώθηση του κανονισμού ευρωπαϊκού του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων. Αναφέρομαι ότι η συζήτηση της σχετικής πρότασης κανονισμού άρχισε κατά την Πολωνική Προεδρία και συνεχίστηκε κατά την Δανική Προεδρία. Η πρόταση συζητήθηκε κατά διάρκεια του Συμβουλίου ΔΕΗ στις 8 Ιουνίου 2012 και αποφασίστηκε ότι το παράρτημα 1, το οποίο περιλαμβάνει τις ουσιαστικές πρόνοιες της πρότασης, θα συζητηθεί στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Επομένως, αν και το θέμα δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες μας, προτιθέμεθα να συνεχίσουμε τη συζήτησή του κατά τη δική μας Προεδρία. Έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν αριθμός αριθμό συναντήσεων της σχετικής ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Όπως όλοι γνωρίζετε, Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέροντο και με σοβαρέ νομικέ προεκτάσει για όλου του εμπλεκόμενου. Είναι το επομένω ότι έχουμε την υποχρέωση ω Προεδρία να δώσουμε σε όλου τον απαιτούμενο χρόνο για να εξετάσουν τι θέσει του γενικά αλλά και ω προ τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις ακούσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Η συζήτηση της πρότασης και ιδιαίτερα του παραρτήματος 1 επιβάλλεται ως εκ τούτου να γίνει με την πρέπουσα λεπτομέρεια, σοβαρότητα και προσοχή. Εξυπακούεται επίσης ότι θα παρακολουθούμε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια στενή και επικοδομητική συνεργασία. Όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα δικαιοσύνη, επισημαίνουμε ότι το Συμβούλιο έχει πετύχει μερική γενική προσέγγιση, ενώ οι διατάξεις για τον οικονομικό φάγελο θα τύχουν διαπραγμάτευση σε οριζόντιο επίπεδο. Για το θέμα αυτό, κρίνοντας από τις μέχρι σήμερα ανεπίσημες επαφές με τους εισηγητές της Επιτροπής Γιούρη και Λίπε, Φαίνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το Συμβούλιο αναφορικά με πολλά κέρια ζητήματα όπως το γεγονός ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των δικαστών το Συμβούλιο ανταποκρινόμενο και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για την κατάρτιση δικαστών έχει αναδείξει το θέμα αυτό το οποίο αποτελεί ένα από τους ειδικότερους στόχους του προγράμματος. Αναντίλεχτα, η κατάκτηση των δικαστών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στην προαγωγή ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πνεύματος και δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους δικαστές, αλλά να επεκτείνεται και στους δικηγόρους, τους δημόσιους κατήγορους και άλλο δικαστικό προσωπικό. Κατά την επιλογή δράσεων προς χρηματοδότηση, η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί τις προτάσεις με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των προτινόμενων δράσεων. Οι δείχτες έχουν αναδιατυπωθεί και διασαφινιστεί, ούτω ώστε να παρέχουν ξεκάθαρη βάση για παρακολούθηση και αξιολόγηση. με βάση τα δεδομένα αυτά, η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο με στόχο την επίτευξη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση μέχρι το τέλος του χρόνου. Τέλος, όσον αφορά θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και ηλεκτρονικού δικαίου, η συνέχιση των εργασιών στον τομέα e-justice κρίνεται ως σημαντική με στόχο τη δημιουργία μιας μονοθυρικής πρόσβασης one-stop shop στον τομέα της δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει ενημερώσει ότι η νομοθετική πρόταση στον τομέα αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2012. Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση. Παρομοίως, η Κυπριακή Προεδρία, στο πλαίσιο των εργασιών όσον αφορά το ήλο, θα συνεχίσει τις εργασίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος όλων των πολιτών. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας για στενή και επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο για επίτευξη του κοινού στόχου της περαιτέρω εδραίωσης ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας προς διευκρίνηση οποιοδήποτε ζητήματος. Σας ευχαριστώ θερμά και εκ μέρους των συναδέλφων ρωτώ τώρα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν έχω σημειώσει κατάλογο. Αλλά παρακαλώ, κύριο Σεύκα, Ταντέους, έχεις το λόγο. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowny panie ministrze. <clears throat> Przede wszystkim Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καταρχάς θα σα ζητήσω θερμά συγγνώμη για την καθυστέρησή μου που οφείλεται σε μια καθυστέρηση στην αύξηση του αεροπλάνου. Ίσως σας φανεί ότι κάποια ερώτησή μου έχει ήδη καλυφθεί από την ομιλία σας και ενδεχομένω να με την άκουσα. Για το κανονισμό Βρυξέλλε 1. Όπως γνωρίζετε, μας απασχολεί πολύ ο τομέας αυτός. Συνεργαζόμαστε ε, με την Προεδρία, είχαμε και με τη Δανική και με την Πολωνική προηγουμένως Προεδρία στενή συνεργασία στο θέμα του κανονισμού Βρυξέλλες 9, μόνο που δεν φτάσαμε στο στόχο μας, στον τελικό στόχο. Δηλαδή σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Και έτσι θα ήθελα να ρωτήσω πώς διαγράφεται το χρονοδιάγραμμα τι σχέδια έχετε για το Συμβούλιο, γιατί βέβαια πάντα έχουμε την ελπίδα να έχουμε τη δυνατότητα να εγκρίνουμε την έκθεσή μας το, φθηνό το φθινόπορο. Μπορείτε να μας δώσετε τις πληροφορίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπερλιγκέρ, παρακαλώ. <clears throat> Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για την εισήγησή σας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για να επαναλάβω την σημασία του κανονισμού Βρυξέλλες 1 που ελπίζουμε να έρθει σε αίσια ο πέρας καθώς και την ε, νομοθεσία σχετικά με την προστασία των θυμάτων καθώς και την πορεία της πρότασης για το δίκαιο των πολίσεων που σίγουρα θα προχωρήσει πιο αργά από τις υπόλοιπες προτάσεις γιατί βρίσκεται σε αρχική φάση αλλά που επίσης έχει μεγάλη σημασία. Θα ήθελα επίσης να, ε, να επιστήσω την προσοχή του Υπουργού στο γεγονός ότι σήμερα συζητάμε σε αυτήν εδώ την ε, ε, συνεδρίαση για ένα σχέδιο πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες για την ε, διαχείριση, τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό και θα θέλαμε να τονίσουμε προς το Συμβούλιο την ε, σημασία αυτής της δραστηριότητας και αυτού του τομέα όπου ακόμα η Κομισιόν δεν έχει δραστηριοποιηθεί, η Εκτελεστική Επιτροπή δηλαδή. Τελευταίο θέμα που θα ήθελα να σας θυμίσω είναι κάτι που με απασχολεί διαρκώς. Είναι το θέμα της κατάρτισης των ε, δικαστών, όπου το επταετές πρόγραμμα, το Justice Program, που προτιθέμεθα να εγκρίνουμε, προβλέπει παρεμβάσεις που μάλιστα έχουν καθοριστεί με πολλαπλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου μας για το θέμα αυτό και γι' αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό και άρα το Συμβούλιο να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα της δημιουργίας μιας ε, νομικής, δικαστικής μάλλον, ευρωπαϊκής δικαστικής νοοτροπίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο Έχουμε εδώ ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχουμε προσδιορίσει μεταξύ των τεσσάρων ε, συνεισηγητών από τις τέσσερις ε, εμπλεκόμενες επιτροπές, Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς, Επιτροπή ε, Νομικών Θεμάτων και έχουμε προβλέψει μέχρι το τέλος ε, του χρόνου ή αρχές του επομένου έτους να είμαστε σε θέση να έχουμε επαληθεύσει όλη την κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε την πρόταση εκθέσεως και άρα στα τέλη της Κυπριακής ή στις αρχές της Ιρλανδικής Προεδρίας θα έχουμε την ε, δυνατότητα να μιλάμε για ενδεχόμενο συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Δεν λέω ότι θα καταλήξουμε αλλά η μητέρα θα είμαστε εμείς από πλευράς μας έτοιμοι να συζητήσουμε για κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν η Κυπριακή Προεδρία θα έχει προχωρήσει αντίστοιχα, αυτή η ερώτησή μου, αντίστοιχα τη δουλειά και γι' αυτό και εγώ ως ένας από τους δύο συνεισηγητές, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Μπερλιγκέρ δεν θα έχει διαφορετική έποψη, ένας από τους δύο συνεισηγητές λοιπόν της Επιτροπής μας, θα ήθελα να πιέσω και να καλέσω να προχωρήσουν αντίστοιχα εργασίες στο Συμβούλιο από πλευρά των ομάδων εργασίας, γιατί είναι αρκετές, δεν είναι μόνο μία, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε παράλληλα και να έχουμε τη δυνατότητα στα τέλη του έτους, αρχές του επομένου μάλλον, ε, υπό την Ιρλανδική Προεδρία να μιλάμε για δυνατότητα συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, είπε ο κύριος Μπερλιγκουερίρ, διότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, έχει πολύ καιρό ε, και πολλή δουλειά πίσω της, αλλά πάντως θα πρέπει Ξέρουμε ότι πρέπει να προχωράμε πάντα βήμα το βήμα, αλλά πιέζουμε, ε, καλούμε μάλλον το Συμβούλιο, παρακαλούμε το Συμβούλιο να εντατικοποιήσει τι εργασίε στο θέμα αυτό. Και δεν βλέπω να ζητεί κανεί άλλο συνάδελφο τον λόγο, γι' αυτό παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τον κανονισμό Βρυξέλλες 1, όπως έχω ήδη αναφέρει Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού, επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο ΔΕΗ των Ιούνιων πολιτική συμφωνία επί του βασικού, επί του βασικού κειμένου της πρότασης, εξαιρουμένων των εντυλογικών σκέψεων και των παραστημάτων. Παρέμεινε να καθοριστεί το ακριβές λεκτικό ορισμένων διατάξεων σε επίπεδο ομάδας εργασίας, καθώς και να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των αιτιολογικών σκέψεων των παραστημάτων. Μετά το τελευταίο Συμβούλιο ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιουνίου συνάντηση ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό. Δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία στα εναπομείναντα σημεία. Συνεπώς η Κυπριακή Προεδρία ανέλαβε να εκπληρώσει την εντολή του Συμβουλίου και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για, να, για τα εναπομείναντα σημεία το συντομότερο δυνατό. Στις 6 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας εργασίας. Το αποτέλεσμα της οποίας θα υποβληθεί προσεχώς στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσωπών και του Συμβουλίου για επιβεβαίωση. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε υπόψη μας και τον προχωρούμε. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε έση εγκατάληξη. Όσον αφορά την εκπαίδευση δικαστών Αναφορικά με το θέμα αυτό, θέλω να επισημάνω ότι είναι πραγματικά τεράστια σημασία της εκπαίδευσης, η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους δικαστές, αλλά να επεκτείνεται και στους δικηγόρους, δημόσιους κατήγορους και άλλων δικαστικών προσωπικών. Χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η εξέλιξη του χώρου δικαιοσύνης και της αμοιβαία εμπιστοσύνης, η οποία αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της αμοιβαία αναγνώρισης. Η θέση αυτή, εξ όσο γνωρίζω, εκφράζει πλήρω και το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο πραγματικά καταβάλει προσπάθειε όπω το όλο θέμα συνεχίσει, συνεχίσει να τοποθετείται ψηλά στην ατζέντα τη Ένωση. Όπω έχω ήδη αναφέρει, στα πλαίσια του πολεετου δημοσιονομικου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-20 και τη πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα δικαιοσύνη, το Συμβούλιο ανταποκρινώνω και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάρτιση δικαστών έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των δικαστών και το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα, τώρα έναν από τους ειδικότερους στόχους του προγράμματος. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συνδράμει τα μέγιστα στην υπερπίδηση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη για χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων. Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για το κοινό Ευρωπαϊκών Δίκαιων των Πολίσεων. Όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Μπερλίγκουε και ο Πρόεδρος, επισημαίνω ότι κατά τις συναντήσεις της ομάδας εργασίας έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις από μεγάλο αριθμό κρατών μελών, αλλά και ενστάσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο προώθησης του ζητήματος και αφορούν μεταξύ άλλων. Πρώτον, την νομική βάση που επικαλείται η Επιτροπή με βάση την συνθήκη. Η θέση της πλειονότητας των κρατών μελών είναι ότι δεν στοιχειοθετείται με βάση τα πραγματικά γεγονότα και τα υπάρχοντα στοιχεία η απαραίτητη ε, αναγκαιότητα που απαιτείται από το άρθρο 114. Δεύτερον, ένας εξίσου σοβαρός λόγος για την ύπαρξη επιφυλάξεων από τα κράτη-μέλη είναι το ότι εφόσον υπάρχουν ήδη άλλα νομικά κείμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδηγίες, που ήδη ρυθμίζουν τα σχετικά ζητήματα, εκτιμάται ότι υπάρχει όχι μόνο επικάλυψη, overlapping, αλλά ότι θα υπάρχει ασυμ, ασυμβατότητα μεταξύ των διαφόρων κειμένων. Συναφώς αναφέρει ότι, ότι σε σχετικό πίνακα αντιστοιχίας τον οποίο ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ύπαρξη επικάλυψης. Πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι μια πλήρης ε, νομοθεσία, ούτε ρυθμίζει απλώς τα τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν, για τα οποία σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει σαφής διατύπωση για την ύπαρξη και έκτασή τους δεδομένου ότι κάποια από τα κείμενα είτε ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια είτε κάποια βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής τους στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επιφυλάξεις εκφράζονται και για τη μορφή του κειμένου. Προτείνεται πρόταση κανονισμού αντί οδηγίας που λόγω της άμεσης εφαρμογής του εκτιμάται ότι μεταξύ άλλων δεν θα είναι συμβατός ούτε με τη Ρώμη 1 για το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε επίσης και με άλλα σχετικά με το ίδιο θέμα κείμενα και διεθνείς συμβάσεις. Με ορατό το ενδεχόμενο να μειωθεί σοβαρά ο φυστάμενος βαθμός προστασίας των οποίων απολαμβάνουν τα αδύναμα μέρη σε μια σύμβαση. Κυρίως γιατί εκτιμάται ότι η προστασία που προβλέπεται στην πρόταση είναι λιγότερη από την προστασία που παρέχεται από άλλα κείμενα, είτε τα τεχνικά δίκαια είτε άλλες διεθνείς νομοθεσίες, έναντι των οποίων ως κανονισμός θα υπερισχύει. Επιφυλάξεις εκφράστηκαν στα πλαίσια της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου και για αρκετά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματο χάρη το πεδίο εφαρμογής καθήλυν, προσωπικό, εδαφικό, τα οποία συζητούνται. Με βάση τα πιο πάνω, είναι προφανές ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί σε τεχνική εξέταση της πρότασης και του παραρτήματος της στο επίπεδο της ομάδας εργασίας πολύ προσεκτικά και διεξοδικά και να δοθεί επαρχής χρόνος στις αντιπροσωπείες να εκφράσουν τις θέσεις τους. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το οποιοδήποτε νομικό εργαλείο σε σχέση με το δίκαιο των πολίσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Όπως έχω αναφέρει και στην αρχική μου τοποθέτηση, θα παρακολουθούμε στενά τις εργασίες, τις εργασίες που προγραμματίζει το Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα αυτό και προσβλέπουμε σε μια καλή και επικοδομητική συνεργασία. Αναφορικά με το θέμα του διοικητικού δικαίου που έθιξε ο κύριος Περλίνγκουερ αυτό είναι, είναι θέμα που τη χάνει χειρισμό από τον Υφυπουργό Προεδρίας για ευρωπαϊκά θέματα, κύριο Μαυρογιάννη και όχι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να, να ρωτήσετε και να πάρετε τις ανάλογες απαντήσεις από τον κύριο και ελπίζουμε να είσαστε και στην Κύπρο οπότε θα συζητηθεί εκτενέστερα αυτό το θέμα. Νομίζω έχω καλύψει όλες τις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Αν παρελπίδα αν έχω φύσικα μια, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Όλοι ευχόμαστε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία για το επόμενο εξάμεινο. Κάθε επιτυχία λοιπόν εξεπλάγει ε, από την απογραφή των προβλημάτων τα οποία παραμένουν ως προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων και η δική μας ανάλυση συμπίπτει βέβαια με αυτήν και πιστεύουμε ότι θα πρέπει και το Συμβούλιο εντατικά να ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο επόμενο εξάμεινο από την Προεδρία σας όπως και εμείς. Ξέρω ότι τώρα πρέπει να πάτε ε, στην Επιτροπή των Εσωτερικών, ξέρω ότι έχουμε θέματα κοινή αρμοδιότητα ε, ω προ το Υπουργείο σα. Σα εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία. Σα ελπίζω για την επόμενη συναντηση. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren. Ξέρετε Εξαιρετούμε κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη προβλέπει παρουσία της Επιτροπής για το σημείο 5 δηλαδή. Δεν έχουν φτάσει όμως ακόμα οι εκπροσωποί Και έτσι πάω στο σημείο 6 για να δώσω το λόγο στην κυρία Νταλόλη, πρόεδρος. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est, c'est Εντάξει, το βρήκα το μικρόφωνο μου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. τα ανοιχτά δεδομένα, open data, είναι γενικές πληροφορίες που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, είτε δωρεάν, είτε για ένα μικρό κόστος. Αυτές οι πληροφορίες στο δημόσιο τομέα αποτελούν μια πρώτη ύλη για προϊόντα και υπηρεσίες με ψηφιακού περιεχομένου και περιλαμβάνουν, ε, μάλλον αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξη για όλα τα κρατημέλη. Η οδηγία 8398 ορίζει ένα, minimum, ένα σύνολο μίνιμουμ κανόνων μεταξύ των οποίων και η διαφάνεια για τη χρήση αυτών των στοιχείων. Το 2011 η Κομισιόν υιοθέτησε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα ανοίγματο δεδομένων που πρέπει να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία με 40 δις ευρώ ετησίως. Ποιες είναι οι βασικές τοποποιήσεις του 2000, του 2003 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Η πρόταση της Κομισιόν ε, εισάγει καταρχήν μια ρητή υποχρέωση για τα κράτη-μέλη ώστε να καταστούν ε, ε, ε, ώστε να δοθεί μάλλον δυνατότητα χρήσης σε όλα τα έγγραφα στα οποία υπάρχει πρόσβαση. Αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσω μιας αδειοδότησης που μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα όσον αφορά το κόστος ε, για τη χρήση αυτών των δεδομένων θα πρέπει να ξεπερνά το μικρό κόστος της αναπαραγωγής και της δημοσίευσης. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, επεκτείνεται στα πολιτιστικά ιδρύματα για όλα τα έγγραφα τα οποία ε, ανήκουν στον δημόσιο τομέα, εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα. Η θέση μου για αυτό το θέμα και ο στόχος μου είναι να προτείνω τροπολογίες που θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες, τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις δημόσιες αρχές να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και να προτείνουν νέες ψηφιακές εφαρμογές. Μάλιστα βρίσκομαι σε μια προοπτική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας και ευκαιριών για νέες θέσεις απασχόλησης, χωρίς φυσικά να ξεχνάμε μια αναυξημένη αποτελεσματικότητα για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε υποχρέωση ψηφιοποίησης όλων των εγγράφων. Η νέα χρήση, η εκ νέου χρήση των δημοσίων πληροφοριών θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο εκτεταμένη. Επιπλέον, θα πρέπει αυτά τα έγγραφα να καταστούν διαθέσιμα σε μορφή που να επιτρέπει εύκολη χρήση των πληροφοριών, χωρίς όμως να προκαθορίζεται ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί. Είναι σημαντικό να ευνοηθεί η χορήγηση ελεύθερων αδειών που επιτρέπουν δηλαδή την τροποποίηση, την αναμετάδοση και την νέα χρήση των ε, λόγω δημοσίων πληροφοριών. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο γιατί αν οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα επιβάλλουν ε, όρους εξαιρετικά αυστηρούς η αγορά δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Δεύτερη παρατήρηση που είναι σημαντική είναι το ύψος των τελών για τη χρήση αυτών των στοιχείων. Είναι προφανές ότι οι αρχές θα πρέπει να, έχουν το... να ανακτήσουν το κόστος που συνδέεται με τη διαδικασία αναπαραγωγής και απάντησης σε ένα αίτημα χρήσης νέας ε, των στοιχείων αυτών. Ωστόσο, τα τέλη αυτά θα πρέπει να οριστούν με σαφή τρόπο, με κάθε διαφάνεια και με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει επίσης να περιορίζονται στα, σε μικρό κόστος γιατί ακόμη μια φορά δημιουργούμε αυτή τη στιγμή μια νέα αγορά. Έπειτα, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα έχει ειδικέ αρμοδιότητες ώστε να εξετάζει τις προσφυγές όσον αφορά την χρήση δημοσίων πληροφοριών. Εδώ είμαι κάπως υποφυλακτική όσον αφορά την δημιουργία και την σκοπιμότητα της δημιουργίας μιας ακόμη ανεξάρτητης αρχής. Έχω την εντύπωση ότι σε κάθε κράτος μέλος μια ήδη υπάρχουσα αρχή θα μπορούσε να αναλάβει αυτές τις ε, αρμοδιότητες βέβαια προς χάρη οικονομίας. Και τέλος, και εδώ είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη για αυτό το θέμα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η νέα χρήση δημοσίων ε, δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα, ορισμένες δημόσιες ε, πληροφορίες μπορεί να αφορούν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, όπως οι ασφαλίσεις, η υγεία τους κτλ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν η απελευθέρωση των δημοσίων ε, δεδομένων έχει, τέτοια φύση που να αποφέρει όλα τα ωφέλη που υπολογίζει η Κομισιόν όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, αλλά σε μια φάση οικονομικής κρίσης και τη στιγμή που η κρίση χρέους δεν επιτρέπει στα κράτη να χρηματοδοτήσουν πολιτικές ανάκαμψης, πιστεύω πως η απελευθέρωση και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα καταθέσω το σχέδιο χνομοδότησής μου μέσα στον Ιούλιο και θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαλό. Δεν βλέπω να είστε κανείς άλλο στο λόγο. Εκ μέρους της Επιτροπής, κύριος Φέτνερ, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας για να ακούσω την πρώτη παρουσίαση από την εισηγήτρια της πρότασής της για αναθεώρηση και βελτίωση της ε, οδηγίας αυτής. Είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις της. σχετικές με τον ε, τομέα το δημόσιο τομέα και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν. Βεβαίως ε, είναι ξεκάθαρες οι ιδέες που υπερασπίζεται η κυρία Γκαλό. Αναφέρεται παραδείγματι στο γεγονός ότι δεν θα πρέπει ένας οργανισμός να υποχρεωθεί να ψηφιοποιηθεί έγγραφα τα οποία δεν ψηφιοποιούνται Συνήθω, προφανώ δεν υπάρχει τέτοιου είδου πρόθεση μέρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασφαλώ θα βοηθάει αν καταστεί αυτό σαφέ, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ω προ την ανεξάρτητη αρχή, αν θεωρείται ότι έχει χρησιμότητα η λειτουργία τη βεβαίω. Ε, διαφορετικά δεν χρειάζεται να θεσπιστεί ένα τελείω καινούριο σώμα, καθώ τα κράτη-μέλη μπορούν την διασφάλιση τη στήριξη των ε, διατάξεων, την υψηλοποίηση δηλαδή της οδηγίας, να την αναθέσουν ωραιότατα σε έναν υφιστάμενο φορέα. Βεβαίω, όπως και η συγγήτρια, έχουμε δεσμευθεί να προστατέψουμε τα απόρριτα δεδομένα, εμπιστευτικά δεδομένα δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Μάσετ, παρακαλώ. Μα ουσίας, αλλά υπάρχει ένα τυπικό που θα έπρεπε να συζητήσουμε. Αφού μας λέει η συγγήτρια πως με την... συνηθισμένη της ε, εξαιρετική ικανότητα θα τα καταφέρει και μέχρι τα τέλη του μηνός θα είναι έτοιμη η έκθεση, θα ήθελα την έκθεση αυτή να την έχουμε αμέσως διαθέσιμη. Δηλαδή, μόλις την καταθέσει να μα στείλει ένα αντίγραφο, ακόμα και αν είναι μόνο στη δική της γλώσσα, για να μπορούμε και εμείς να εργαστούμε στους ίδιους ρυθμού που εργάζεται και η ίδια, που επαναλαμβάνω είναι εξαιρετικά γρήγορη. Και βεβαίω μόλις ε, διατυπωθεί η έκθεση θα την δείτε και γραπτό. Ας περάσουμε τώρα πάλι στο σημείο 5, μια και έχουμε εδώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής για το Πεκίνο, εάν είναι έτοιμη. Η κυρία Μαρία Μάρτιν Πρόψη, είστε εδώ πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και στο συγγνώμη που χρειάστηκε η Επιτροπή σας ε, να περιμένει. Είχαμε ενημερωθεί ότι θα συζητηθεί για τις 4 το θέμα αυτό στην Επιτροπή σας και γι' αυτό είχαμε αυτή τη μικρή διαφορά. Είμαι εδώ λοιπόν για να ενημερώσω απλώς την Επιτροπή σας για την ε, σύναψη στην, ε, στο Πεκίνο σε μια διπλωματική διάσκεψη που έλαβε εκεί η χώρα και ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουνίου ε, την προηγούμενη εβδομάδα μιας νέας διεθνούς συνθήκης για την προστασία των οπτικοακουστικών του οπτικοακουστικού υλικού. Πρόκειται για την συνθήκη οπτικοακουστικών επιδόσεων. Ουσιαστικά προς στόχο έχει να προστατεύει τους ηθοποιούς αλλά βεβαίως και μουσικούς ή όποιον άλλον ερμηνευτή που παρουσιάζεται μέσα σε οπτικοακουστικό υλικό. Είτε πρόκειται για ταινία, είτε πρόκειται για μουσικό έργο, τηλεοπτική ταινία ή σειρά, ε, ντοκιμαντέρ. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό και γιατί γίνεται τώρα. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία τράβηξε σε χρόνο αρκετά. Είναι νομίζω μια από τις λίγες περιπτώσεις όπου διπλωματική διάσκεψη κράτησε 12 ολόκληρα χρόνια. Η διπλωματική διάσκεψη άρχισε και ολοκλήρωσε το από το έργο της ε, το 2000, μέσα στο έτος του 2000, μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή είχε τελειώσει τα θέματα, αλλά το, στο σημείο αυτό το χρονικό και και ότι υπήρχε ήδη συμφωνία επί των περισσότερων άρθρων της συνθήκης, που θα εξασφάλισαν δικαιώματα για τους ε, ηθοποιούς, προέκυψε διαφωνία εντονότατη για ένα μόνο άρθρο, το άρθρο το οποίο έχει να κάνει με την εκχώρηση δικαιωμάτων από τον ερμηνευτή, ερμηνευτή στον παραγωγό. Και για να εξηγήσω για όσους είναι κάπως πιο εξοικειωμένοι με τον τομέα των, ε, τηλεπικοινωνιών, των οπτικοακουστικών, πρόκειται για ένα ζήτημα ακανθόδες για πολλές χώρες στον κόσμο. Υπάρχουν διαφορετικέ λύσεις. Το 2000 έγινε εντονότατη αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείες θέλησαν να, να επιβάλλουν τη δική τους οπτική, το δικό του σύστημα δηλαδή, την αυτόματη εκχώρηση των δικαιωμάτων του ε, ηθοποιού στον παραγωγό της ταινία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια πιο ευέλικτη, πολύ πιο ευέλικτη προσέγγιση, καθώς στα κράτη-μέλη επικρατούν διαφορετικές λύσεις. Χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία έχουν διαφορετικά συστήματα από αυτά της Ισπανίας, του Βελγίου ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή ήταν και η υπόθεση, αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο ε, σταμάτησε τις εργασίες σε αυτή τη διπλωματική ε, διάσκεψη χωρίς να τελειώσει. Παρέμεινε εκρεμές λοιπόν το θέμα για μια δεκαετία και μόνο στα τέλη του 2011 κατέστησε σαφές ότι υπήρχε η δυνατότητα να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Δηλαδή να συνάψουμε τη συνθήκη στη μορφή που είχε ήδη το 2010 προσλάβει και να προσθέσουμε και ένα άρθρο, το υπαριθμών 12 τώρα της συνθήκης, για την εκχώρηση των δικαιωμάτων, το οποίο αφήνει απόλυτη ευελιξία για τα συμβαλόμενα μέρη και έτσι αυτά μπορούν να διατηρήσουν τα συστήματα που έχουν ως προς την εκχώρηση των δικαιωμάτων. Ε, αυτή λοιπόν η συναντήληψη, η αντίληψη δηλαδή από πλευρά των ΗΠΑ ότι μπορούν να δεχθούν το δικό του σύστημα, να διατηρήσουν το δικό του σύστημα χωρί να το επιβάλλουν στου άλλου συμβαλωμένου και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν τα διάφορα κράτη να κρατούν στα δικά του συστήματα. Αυτή η ευελιξία λοιπόν η οποία αντικατοπτρίζεται στη συνθήκη κατέστησε δυνατή την ε, ανάληψη των εργασιών στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής διάσκεψης στο ε, Πεκίνο και την σύναψη της συνθήκης που επιτύχαμε τώρα. Έχουμε λοιπόν σαν αποτέλεσμα μια, ένα αυξημένο επίπεδο προστασίας για τον ηθοποιό, για τον ερμηνευτή ε, και στο πλαίσιο του περιβάλλοντος ίντερνετ, του διαδικτύου, πράγμα το οποίο είχε γίνει για τους ε, παραγωγούς ε, καταγραφής φωνής, για τους ηθοποιούς και τα σε μια αντίστοιχη συνθήκη του 96 ο ηθοποιός δεν είχε καλυφθεί, καλυπτεί, καλυφθεί προς την προστασία στο διαδίκτυο των δικαιωμάτων του και ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό ότι ο ερμηνευτής στον τομέα των οπτικοακουστικών έχει στην Ευρώπη βέβαια ήδη υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας και τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει η συνθήκη ήδη καλύπτονται αντικατοπτρίζοντας τις υφιστάμενες οδηγίες ειδικότερα την οδηγία του 1992 που ορίζει τα ε, βασικά δικαιώματα σχετικά με την ε, ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού και την μεταγενέστερη οδηγία για το διαδίκτυο. Άρα εδώ αυτή η συνθήκη έχει σημασία ε, για, την περίπτωση όπου ο ηθοποιός έχει ή το προϊόν του ηθοποιού έχει την χάνει εκμετάλλευση σε τρίτες χώρες και μην, σκέφτεστε μόνο την περίπτωση μιας ταινίας ε, κινηματογραφικής αλλά και βέβαια τις ταινίε τις τηλεοπτικές ή τις σειρές οι οποίες έχουν μεγάλη διαδοσία ανά τον κόσμο και ως εκ τούτου ε, ο ηθοποιός ε, που έχει παίξει σε μια τέτοια σειρά εφόσον αυτή ε, πολιθεί στο εξωτερικό θα έχει αυξημένη προστασία δυνάμει της συνθήκης που συνήφθη. Τώρα αυτή είναι με αδρές γραμμές η περιγραφή των κυρίων πλέον εκτιμάτων που προσφέρει αυτή η νέα συνθήκη. Πότε θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη. Χρειάζεται 30 συμβαλόμενα μέρη να την ε, κυρώσουν. Άρα θα περάσει κάποιο διάστημα, ασφαλώς. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει από πλευρά τη να ξεκινήσει η διαδικασία καταρχά βέβαια τη υπογραφή, που είναι το πιο τυπικό, ε, η πιο τυπική φάση για την αναγνώριση συνθήκη, αλλά ταυτόχρονα και την ε, συμφωνία από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Συμβούλιο βασικά και το Κοινοβούλιο, να κυρωθεί η συνθήκη. Αυτή είναι η προσπάθεια στην οποία θα, θα από, το, από τώρα και ιδιαίτερα το φθινόπωρο, συστούμε με εσά, συστούμε με τα κράτη-μέλη και επισημαίνουμε ότι δεν χρειάζεται τροποποίηση τη υφιστάμενης ευρωπαϊκή επίπεδο νομοθεσία, δεν χρειάζεται ούτε αναθεώρηση ούτε νέα νομοθεσία δεν υπάρχουν θέματα τα οποία να βρίσκονται εκτός του ευρωπαϊκού κεκτημένου ή όποια είναι δεν χρειάζονται εναρμόνιση και έτσι εν αυτή την ενία το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι μια συνθήκη η οποία έπρεπε να έχει συναυθεί πριν από 10 χρόνια τώρα την έχουμε βάσει περιπτώσει αλλά πάντως ε, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους ε, ερμηνευτές ανά τον κόσμο, τις ε, εταιρείε ε, ίσπραξης δικαιωμάτων που τους εκπροσωπούν, αλλά βέβαια και τους παραγωγούς. Και βεβαίως με στη θέση σας, αν τυχόν θέλετε να συστήσουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν ερωτήσεις από πλευρά των συναδέλφων. Ο κύριος Μάσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα στηρίξω και θα στηρίξω με ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία για τη συμφωνία αυτή και οι εξηγήσει που ακούσαμε σήμερα ήταν πολύ ικανοποιητικέ γιατί θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει και το χώρο και την ηθοποιία και τη σημασία που έχουν. Ζούμε σε ένα κόσμο από τότε που ο Ντάριο Φω πήρε το Νόμπελ που θα ήταν αφάνταστο το ότι θα μπορούσαμε να βιώσουμε μια τέτοια στιγμή όπου οι επιθυμίες του δημιουργού θα προστατεύονται με τέτοιο τρόπο. Ξέρουμε τι κάνει η ΕΜΚΟ και ξέρουμε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε όταν θα περάσει ε, αυτό το θέμα από το Κοινοβούλιο. Και οι συγγραφείς και οι ηθοποιοί αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Μετά το καλοκαίρι και ακολουθώντας και το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση από τις ε, κοινοτικές αρχές, ε, αναρωτιέμαι τι πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, πότε θα μπορέσουμε εμείς να δώσουμε την τελική έγκριση. Γιατί φοβάμαι ότι θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ, όπως συμβαίνει συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ ε, για την παρουσίασή σας. Θα είχα να κάνω την εξή ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα περίφθη η πρόταση άκτα από την ε, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. και θα ήθελα να ρωτήσω η πρόοδος ως προς την σύναψη της εν λόγω συμφωνίας διαφέρει από αυτήν, από τη διαδικασία δηλαδή, που ακολουθήθηκε για την άκτα πρώτον και δεύτερον μπορείτε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες ως προς την ε, σωστή αμοιβή για, τη, για τα δικαιώματα αυτά των ερμηνευτών. Μπορείτε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες. Και ο πρόεδρος, αν μου επιτρέπετε, μια προκλητική ερώτηση. Υπάρχουν ήδη, ακούγονται ήδη φωνές ε, ίσως ε, για ε, απειλές κατά της ελευθερίας ε, στο διαδίκτυο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις, ακόμα και τις πιο προκλητικές. Να τις απαντήσω με τη σειρά που έγιναν. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα. Για να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη χρειάζεται 30 επικυρώσεις και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικυρωθεί από τα 27 κράτη-μέλη 28 κράτη-μέλη από το χρόνο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είμαστε σε αρμοδιότητα κοινοτική αλλά και εναρμόνιση σε εθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν θα πρέπει, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συγχωρείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διορθώνω να επικυρώσει όπως θα κάνουν και τα κράτη-μέλη. Τι έχουμε κάνει στην πράξη στο παρελθόν. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ε, επαναλάβουμε, αλλά θα περιμένουμε να έχει τελειώσει η επικύρωση από τους υπόλοιπους και θα επικυρώσουμε όλοι μαζί καταθέτοντας το ε, κείμενο της επικύρωσης ε, στη Γενέβη. Μαζί, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει στα κράτη-μέλη, αλλά συνήθως έτσι κάνουμε. Για το χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος μπορεί παραπάνω. Γιατί χρειάζεται να επικυρωθεί και από τα 27 κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε καταλαβαίνετε πως οι διαδικασίες αυτές αργούν. Για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των διαπραγματεύσεων και των διαπραγματεύσεων για την άκτα, νομίζω πως ε, το πολύ θετικό αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε περάσει σε ανοιχτές και πολύπλευρες σχέσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων, ο WIPO, συνήθως εγκρίνει συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι η Σύμβαση Ρώμης και είναι όλοι οι συμβάσεις ε, του 1996 και η σημερινή που έχουν ε, υπογραφεί εκεί με συμμετοχή πάνω από 150 κράτη, το οποίο ήταν παρόντα στο Πεκίνο, ήταν παρόντα και το 2000 στη Γενέβη, όλα τα κράτη αυτά και σημαίνει ότι έχουμε και συμμετοχή διακυβερνητικών οργανώσεων και βέβαια είναι διαπιστευμένες και ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στον WIPO. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για, την, για να υπηρετήσουμε τη διαφάνεια και βάσει της εντολής που είχε δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε, ακολουθήσαμε ακολουθήσαμε μια τελείως διαφορετική διαδικασία από αυτή που είχαμε για την άκτα. Uh, the remuneration rights, uh, indeed, this is an issue that... Για τα διάφορα τέλη, για τους ερμηνευτές προστατεύονται. Προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση το κεκτημένο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. Και είμαι σίγουρη πως οι συζητήσεις αυτές θα μας οδηγήσουν στο να αξιολογήσουμε κατά πώς είναι αρκετό να έχουμε κάποια αποκλειστικά δικαιώματα ή αν χρειάζεται να αναγνωρίσουμε επίσης και το δικαίωμα στις αμοιβέ. Ε, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν δίνουμε την ευκαιρία στους μουσικούς, τους ηθοποιούς, στους χορευτές οι οποίοι παρουσιάζουν σε κάποιο όπτικο ακουστικό μέσο να έχουν τη δυνατότητα να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις όλο τον κόσμο πως έχουν δικαιώματα και αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Τώρα για την ερώτηση που κάνετε για το με ποιον τρόπο τα δικαιώματα αυτά θα δημιουργήσουν πρόβλημα για την ελευθερία έκφρασης και την λειτουργία του ίντερνετ του διαδικτύου. Δεν θα σας εκπλήξω αν σας πω πως την αξιολόγηση που κάναμε δεν θα έχει καμία επίπτωση υπάρχει το θεμελιώδες δικαίωμα των δικαίωμα των ερμηνευτών που μας δίνουν την ώρα τους και το ταλέντο τους και τη δημιουργικότητά τους και ε, φτιάχνουν αυτά τα, τις ταινίε και τα έργα τα οποία ε, όλοι θέλουμε να παρακολουθούμε να αμείβονται. Και δεν μιλάμε μόνο για μεγάλους Αμερικάνους και Ευρωπαίους στάρ, μιλάμε για πάρα πολλούς ερμηνευτές Χωρίς αυτούς δεν θα βλέπαμε ούτε ταινίε, ούτε θα είχαμε τον ε, κλάδο των οπτικοακουστικών ε, στην Ευρώπη που όλοι τόσο απολαμβάνουμε. Για να σας δώσω και την τελική απογραφή των κρατών που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συνθήκη αυτή, ναι, η ΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και άλλους που θα πρέπει να μην ξεχάσουμε γιατί αποδεικνύει αυτό πως πολύ ενδιαφέρονται για τα οπτικοακουστικά σε διάφορα κράτη, σε, άλλα, σε άλλες φάσεις ανάπτυξης. Βραζιλία, Ινδία. Η Ινδία είναι πολύ μεγάλος παραγωγός οπτικοκουστικών έργων. Νιγηρία και Σενεγάλη, για παράδειγμα, στην Αφρική. Πολύ θετικό λοιπόν πως για πρώτη φορά έχουμε τέτοιου είδους ε, συνθήκη για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρει το όνομα χώρας η οποία είναι ακόμα αναπτυσσόμενη. Έχουμε τη σύμβαση της Βέρνης, της Γενέβης και τώρα έχουμε και αυτή του Πεκίνου. Για να αναγνωρίσουμε και να προστατεύσουμε εδώ τους ηθοποιούς, κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα σε ποια φάση ε, ανάπτυξης βρίσκονται αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, πληρέστατη απάντηση στις απαντήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια το εγχείρημα, το οποίο Περιμένουμε να δούμε κι εμείς. Στο 34, τον κύριο Λεμπερνικουέρ τώρα θα ακούσουμε για το διοικητικό δίκαιο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας όταν εγκρίναμε το έγγραφο εργασίας στις 21 Νοεμβρίου οποίο <clears throat> οδήγησε στη σύνταξη αυτής της έκθεση πρωτοβουλία Πρόκειται για ένα νέο θέμα, νέα ύλη για την Επιτροπή μας και για την Ευρώπη. Θέλω να υπογραμμίσω την ε, καινοτομία διότι πρόκειται για κάτι για το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε ιδιαίτερα, αλλά σηματοδοτεί και ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την Ευρώπη που παραδοσιακά το διοικητικό δίκαιο ήταν αρμοδιότητα των κρατών. Η Ευρώπη επιμένει δεν θέλει να είναι κράτος, αλλά ε, πρέπει να δει ποια είναι η πραγματικότητα, η διοικητική που πια έχει διευρυνθεί και άρα υποχρεούται να ορίσει διοικητικά ε, τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και διοικητικού μηχανισμού, προσωπικού που εργάζεται, με ένα κράτος, που εργάζεται για ένα κράτος και ε, έχει επαφές με το κράτος αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως η Ευρώπη έχει γίνει κράτος, αλλά ήδη διαβάσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες ότι η ευρωπαϊκή πολιτική οντότητα θα μπορούσε να ορίζεται μέσω του καθορισμού των πολιτικών δικαιωμάτων των ε, πολιτών της Ένωσης απέναντι στην διοίκηση, στο διοικητικό μηχανισμό αυτής της ίδιας. Άρα λοιπόν όχι μόνο θα ενισχυθεί η νομιμότητα της Ένωσης, αλλά και θα δοθεί ένα σαφής καθορισμός των προσδοκιών και των δικαιωμάτων των πολιτών που πρέπει να αποσαφενιστούν περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα και έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια μεγαλύτερη βεβαιότητα δικαίου όταν θέλουμε να ορίσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες και την διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να πω ότι η πολιτική πρόταση που κάνουμε εμεί σήμερα πέρα από τη λειτουργία και την ε, πρωτοβουλία που προτείνεται από, την, από μας Η πρωτοβουλία αυτή βασικά στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να κάνει το καθήκον της, να αναλάβει την πρωτοβουλία για να υποβάλει μία πρόταση κανονισμού που αφορά την διοικητικές διαδικασίες. Και θα ήθελα να το πω αυτό όχι μόνο για ε, ακαδημαϊκούς λόγους αλλά και γιατί σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γιούρη ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Σεύκοβιτς νομίζω ήταν αντιπρόεδρος που είναι και συναρμόδιος για τέτοια θέματα ενώ του ζητήθηκε να, κάνει, να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα ε, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έκανε αυτή την αρχική μας εργασία η οποία μας οδήγησε σε αυτό εδώ το σημερινό κείμενο ε, μάλλον θα ασχολείται με αυτό το θέμα σαν να ήταν μια όριστη δραστηριότητα σαν να μας ενδιαφέρει. η δηλαδή κάποιες αφηρημένες αόριστες λύσεις, ενώ η Επιτροπή, ε, η οποία είναι το εκτελεστικό όργανο, ε, ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Με σε αυτού του είδους η προσέγγιση και εμείς θέλουμε να ε, καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ίσως να έχει μεγαλύτερη αίσθηση του συγκεκριμένων θεμάτων, να κάνει το καθήκον της και να παρουσιάζει μια νομοθετική πρωτοβουλία σε σχέση με τον πολιτική πειθαρχία ε, για όλες αυτές τις διαδικασίες. Εμείς ε, θέλουμε θέλαμε, το θέμα το οποίο μας απασχολεί να αφορούσε μόνο τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι δηλαδή τα μονομένα κράτη, όχι, όχι τις ε, διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, γιατί αυτά δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας, αλλά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τομέων παρέμβασής της. ώστε να ε, περιοριζόμαστε σε έναν πυρήνα γενικών κανόνων και να δημιουργηθεί έτσι ένας de minimis κανόνας εκεί όπου δεν υπάρχει λέξη specialis, ειδικός, ειδική δηλαδή σχετική νομοθεσία. Και να μην μπούμε σε εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες, αλλά να υπάρχει ωστόσο ένα σημείο αναφοράς ώστε να κωδικοποιηθεί ένας πυρήνας γενικών αρχών για την χρηστή διαχείριση με έναν ελάχιστο αριθμό διαδικαστικών κανόνων που θα ορίζουν τα καθήκοντα διαφάνειας και υπευθυνότητας στη διαχείριση της διοίκησης και έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα δικαίου και να γίνονται σεβαστές, σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη διοίκηση. Σήμερα υπάρχει το άρθρο 41 των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει συμπεριληφθεί στη συνθήκη και άρα είναι ισχύων κανόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου γίνεται λόγος για το ευρωπαϊκό δίκαιο και για την ε, χρηστή, μάλλον τον, έναν κώδικα διοντολογίας για το διοικητικό μηχανισμό. Έχουμε δηλαδή νομική βάση. Έχουμε εμπνευστεί αυτές τις ιδέες και από τις αρχές που διεύουν ε, τον κώδικα διοντολογίας ε, της διοίκησης ε, από την νομολογία του 10. Αυτή είναι η φιλοσοφία η νομικοπολιτική η οποία επηρέασε την πρόταση που εγώ σας υποβάλλω και δεν θα σας υποβάλλω σε λεπτομερή παρουσίαση των των ε, διατάξεων που προτείνουμε για τις σχέσεις δηλαδή μεταξύ των γενικών κανόνων και των ε, το, τομεακών μέσων και των αρχών που θα πρέπει να διέπουν όλες αυτές τους κανόνες που είναι βασικές αρχές του διοικητικού ε, δικαίου όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν ε, τις αποφάσεις που υιοθετεί η διοίκηση και ούτω καθεξής, όσον αφορά την αναθεώρηση και τη διόρθωση διοικητικών αποφάσεων, τη μορφή του κανονισμού και τη δημοσίευσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Δεν είστε κανεί άλλο το λόγο. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Σα ευχαριστώ θερμά για τη δουλειά που κάνατε εδώ. Πρέπει να προσδορίσουμε προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 19 Σεπτεμβρίου, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Και τώρα περνάμε στη συνεδρίαση κλεισμένων των θυρών. Διακόπτω για λίγο και όποιος δεν έχει θέση εδώ παρακαλώ να αποχωρήσει και παρακαλώ να βγούμε και offline για να μην μεταδιδόμαστε πλέον στο διαδικτύο. Okay.